πρακτικό και τα εγκεκριμένα κείμενα της ε, περίοδου συνόδου 4 Φεβρουαρίου 2016 είναι διαθέσιμα, υπάρχουν ενστάσεις. Ρωτώ. Όχι. Θεωρώ λοιπόν ότι το πρακτικό εγκρίνεται. Α, με συγχωρείτε, κυρία Φλάνναγκαν για το πρακτικό. Α, με συγχωρείτε, ο κύριος Uh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιθυμώ να κάνω μια προσωπική δήλωση. Στην τετάρτη της συνόδου του Στρασβούργου έλαβα το λόγο και ρώτησα τον κύριο Γιούνκερ, του υπέβαλα ερώτηση για το πρόβλημα των τραπεζών στην Ιρλανδία. Είχα ελπίσει ότι μιλούσα σε περιβάλλον που θα έχερα την προστασία του Προεδρείου. Ωστόσο, όταν τα πρόσωπα του γραφείου μου εξέτασαν το βίντεο μετά από την συνεδρίαση, άκουσαν τον πρόεδρο που είχε ξεχάσει το μικρόφωνο του ανοιχτό να εκφωνεί Jesus Christ. Ίσως επειδή έχω μακριά μαλλιά και γέννη ή μήπως δεν του άρεσαν τα όσα λέω. Δεν με ενδιαφέρει ωστόσο αν ο πρόεδρος του αρέσουν ή δεν του αρέσουν αυτά που λέω. Η δουλειά του είναι να είναι ουδέτερος και ανεξάρτητος. Αν θέλει να κάνει πραγματικά τη δουλειά του, αντί να απελπίζεται για αυτά που λέω εγώ και που δεν του αρέσουν, καλύτερα να φροντίσει να απαντήσει ο κύριος Γιούνκερ. Επιθυμώ λοιπόν να ακούσω συγγνώμη και στο όνομα των ανθρώπων που με έχουν ψηφίσει και με έχουν αποστείλει εδώ, διότι είναι προσβλητικό να ακούσω τέτοια φράση σε βάρος μου ή να πει κάποιος κάτι τέτοιο μόλις κάποιος όπως εγώ έχει τελειώσει την δήλωσή του. Αν λοιπόν ο άνθρωπος αυτός επιθυμεί να αποδείξει ότι είναι ανεξάρτητος, διότι δεν μου φαίνεται εδώ στο Προεδρείο να υπάρχουν και πολλοί ανεξάρτητοι, μπορούν να αποδείξουν ότι είναι. Zunächst hat sich äh, Επί του σημείου αυτού έχει ζητήσει το λόγο ο Αντιπρόεδρος κ. Λάμπστορφ. Όχι. Καλά, καλά. Όχι, μου λένε ότι ο κύριος Λάμστορφ προείδρευε το χρονικό εκείνο σημείο όπου σας χαρακτήρισε ως Ιησού Χριστό. Ε, θα το εξετάσουμε κύριε συνάδελφε και θα επανέλθω να σχολιάσω την παρέμβασή σας. Ο κύριος Πάσκου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιθυμώ να ενημερώσω το σώμα για ένα θέμα ελευθερίας εκφράσεως στη Ρουμανία. Προετών διοκτήτη πέντε τηλεοπτικών σταθμών, δύο ραδιοφωνικών σταθμών και δύο εφημερίδων καταδικάστηκε σε δεκαετή φυλάκιση. Συνεπώς και τα περιουσιακά του στοιχεία δημεύτηκαν. Προ λίγων ημερών οι φορολογικές αρχές πήγαν στα γραφεία του ΙΝΤΕΚ της ε, ε, ε, εταιρείας αυτής για να την εξώσουν. Ωστόσο, δεν έχουν καμία σχέση οι ε, άνθρωποι της εταιρείας Συντάκ με το θέμα αυτό. Εγώ θεωρώ την κίνηση αυτή απαράδεκτη. Κοιτάξτε κύριε Πασκού, είστε αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οφείλετε να γνωρίζετε ότι αυτό το θέμα δεν εντάσσεται στην ημερήσια διάταξη. Μπορείτε να κάνετε τη δήλωσή σας αυτή σε κάποιο άλλο χρονικό σημείο. Και θα επιτρέψω μόνο πλέον την τη λήψη του λόγου συγγνώμη, για θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ναι, κύριε Άντερσον, μόνο όμω για θέμα ημερησία διατάξεω ή συγκεκριμένο διαδικαστικό αίτημα. Γνωρίζω ότι στην Ιρλανδία διεξάγεται προεκλογική εκστρατεία. Αλλά εκεί δεν μπορώ να σα βοηθήσω και περισσότερο. Ίσως θα... θα ζητήσετε συγγνώμη όταν ακούσετε τι θέλω να πω. Επιθυμώ να εφιστήσω την προσοχή σας και της Αντιπροέδρου κυρίας Μογκερίνη σε έναν απεργό πείνας, Παλαιστίνιο, 33 χρονών, δημοσιογράφο, πατέρα δύο παιδιών, που διεξάγει η απεργία πείνας επί 92 ημέρες. Άνθρωπος ο οποίος κρατείται χωρίς δίκη, χωρίς απαγγελία κατηγοριών. Πεθαίνει ο άνθρωπος αυτός. Ο γιατρός λέει ότι είναι στο χείλος του θανάτου. Απευθύνουμε έκκληση στην Αντιπρόεδρο Μογκερίνη να παρέμβει Μιλήστε μαζί της. Μιλήστε και σώστε τη ζωή του ανθρώπου αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρος. Ανακοινώσεις.